Euh, Θα συμφωνήσετε λοιπόν με αυτές τις αλλαγές. Θα ήθελα να σας ενημερώσω για το εξή τώρα. Η Επιτροπή των Προϋπολογισμών και η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων ως συναρμόδιες επιτροπές επί της ουσίας ε, βάσει του άρθρου 55 του κανονισμού η Επιτροπή Μεταφορών Τουρισμού ε, και Ήτρε επίσης βάσει του άρθρου 54 του κανονισμού. Αυτές οι δύο θα επιληφθούν διότι στους ζητήθηκε στις 21 ε, Αυγούστου ε, βάσει ε, του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2015-2017 για να δημιουργήσουν ένα βαθμολόγιο ή ένα πίνακα δικτών ε, στα πλαίσια των στρατηγικών επενδύσεων έτσι ώστε να υπάρξει μια ανεξάρτητη αξιολόγηση όσο και διαφανής για τη χρήση της εγγύησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πάρα πολύ ε, σύντομη η προθεσμία αντίρρησης και εκτάκτος. Στις 30 του μηνός Ιουλίου σας διαβιβάστηκε το αίτημα και μέχρι τις 31 Αυγούστου δεν υποβλήθηκε στη γραμματεία της Επιτροπής μας καμία ένσταση ή αντίρρηση. Οπότε όπως ορίζει το άρθρο 23 παράγραφος 5 του Κανονισμού Ευρωπαϊκή Ένωση 2015 κάθετος 2017 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Ισχύουν ε, λοιπόν ε, οι διατάξεις αυτές και σας παραπέμπω επίσης στο άρθρο 105 και 107 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως προς αυτό. Έχετε λάβει το σχέδιο των πρακτικών των συνεδριάσεων της 15ης και 16ης Ιουλίου. Έχετε σχόλια, παρατηρήσεις, άρα μπορούν να θεωρηθούν εγκεκριμένα τα εν λόγω πρακτικά. Εγκρίνονται τα πρακτικά. Λοιπόν, θα παρακαλέσω τώρα τον εισηγητή μας, τον γενικό εισηγητή και τον εισηγητή για τα λοιπά τμήματα να μας ενημερώσουν για την κατάσταση όπως έχει στις παραμονές της θέσης ε, του Συμβουλίου, του Κορεπέρ δηλαδή, για το σχέδιο προϋπολογισμού 2016. Αγαπητέ Φερνάντες. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και θα ήθελα να καλωσορίσω και όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους για το θέμα αυτό το οποίο στην Επιτροπή μας ε, και στο Κοινοβούλιο και στην Ολομέλεια έχει εκτεταμένως συζητηθεί. Έχουμε δύο ψηφίσματα από το Κοινοβούλιο. Στο πρώτο ψήφισμα αναφέρονται οι κατευθυντήριες γραμμές, οι προτεραιότητες οι οποίες ορίζουμε για την απασχόληση, για τις μικρομεσαίες και τις ε, πολύ μικρές ε, επιχειρήσεις, για την επιχειρηματικότητα, για την αλληλεγγύη, την εσωτερική και την εξωτερική, επικεντρωνόμενη στο θέμα της μετανάστευσης. Με απότερο στόχο να μπορέσουμε να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις ε, τις οποίες έχουμε αναλάβει, με τον σκοπό τον οποίο έχουμε ορίσει στο χρηματοοικονομικό στο σχέδιο προπολογισμού. Έχουμε λοιπόν σαφέστατε προτεραιότητες, προτεραιότητε, οι οποίε ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, μπορούμε να πούμε ότι υποστηρίζονται από την ευρεία πλειοψηφία για τα συγκεκριμένα θέματα τώρα των προτεραιοτήτων. Δεν ε, μπορούμε να αποφύγουμε και φυσικά δεν μπορώ παρά να τονίσω το πόσο επίγον είναι το θέμα τη μετανάστευση και των προσφύγων. Ήδη από τι αρχέ του έτου το Κοινοβούλιο έχει κινητοποιηθεί για την προτεραιότητα αυτή. Είναι πραγματικά απαράδεκτο και είναι αδιανόητο το πώ τοποθετείται το Συμβούλιο για τι περικοπέ ε, που γίνονται στο τομέα αυτό. Το Συμβούλιο λοιπόν επεξηγεί και ε, δικαιολογεί τις προθέσεις και στην πράξη ουσιαστικά τι κάνει περικοπές σε τομείς όπου το Κοινοβούλιο είναι στεναρό, όπου είναι στεναρική στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τι να φανταστεί και ο πολίτης, λοιπόν. Δεν υπάρχει Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. και στο θέμα των προσφύγων της ε, μετανάστευσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε προτάσεις, αλλά το Συμβούλιο δεν μπορεί να αποφασίσει ποια κοινή πολιτική θα ακολουθήσει και ακόμα χειρότερο κάνει περικοπές. Περικοπές σε εργαλεία, σε μέσα που αφορούν την μετανάστευση. Το θέμα λοιπόν είναι το εξή. Τι προτίθεται να κάνει το Συμβούλιο, τι θέλει να κάνει το Συμβούλιο, δεδομένου και του έκτακτου χαρακτήρα η απάντηση είναι ότι δεν κάνει προσπάθειες. Αντιθέτως, θέλει να περικόψει και αυτά που ήδη προβλέπονταν στο ετήσιο πρόγραμμα βάσει των, ε, του πολιτούς ε, προγράμματος. Για παράδειγμα, στην ε, τμήμα 4 προτείνονται περικοπές στις υποχρεώσεις πληρωμών. 163 εκατομμύρια Πώς να το δεχτούμε λοιπόν αυτό. Ότι γίνονται δηλαδή περικοπές, 75 εκατομμύρια στις υποχρεώσεις, στα εργαλεία για την ε, ε βοήθεια. Όλα αυτά λοιπόν πώς μπορούμε να τα αποδεχτούμε. Το Συμβούλιο λοιπόν ε, θέλει να κάνει περικόπες 39,8 εκατομμύρια στις ε, ε, δεσμεύσεις, 143 εκατομμύρια στις πληρωμές. Είναι εντελώς αντίθετη λοιπόν και αντιφατική. Υπάρχει μεγάλη αντίφαση μεταξύ του τι λένε και του τι κάνουν τελικά. Περικόπτουν τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και πληρίζουν τη φιλοδοξία του προϋπολογισμού. σε ό,τι αφορά το Κοινοβούλιο τώρα, σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη προτεραιότητα. Πάντα ήμασταν υπέρμαχοι του κοινοτικού κεκτημένου, των κοινοτικών αξιών, της αλληλεγγύης, της ανθρώπινης ε, αξιοπρέπειας. Πολύ απλά λοιπόν δεν μπορούμε να αποδεχτούμε αυτή την αδιαφορία από πλευρά του, του Συμβουλίου. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε το γεγονός ότι δεν υπάρχει κοινή πολιτική, ότι δεν υπάρχει δράση, ότι δεν υπάρχει επαρκή χρηματοδότηση από πλευρά του Συμβουλίου. Το πρόβλημα λοιπόν είναι στο Συμβούλιο. Βλέπουμε να επικρατεί τελικά τα, η εθνική συμφεροντολογία και οι εθνικοί εγωισμοί. Τα κράτη-μέλη ζητούν ε, αλληλεγγύη μέσω του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Οι χώρες που λαμβάνουν δηλαδή τους πόρους ε, από τα μία συνοχής, από τα διευθυντικά ταμεία. Οι χώρες όμως αυτές δεν μπορούν να επιδείξουν οι ίδιες ε, αλληλεγγύη σε τα θέματα αυτά. Η αλληλεγγύη είναι αμφίδρομο σύστημα, ξέρετε. Δεν μπορούμε μόνο να παίρνουμε και να μην είμαστε διτεθειμένοι να δίνουμε το οτιδήποτε. Είναι θέμα δούνα και λαβή. Ας δούμε λοιπόν και τις άλλες προτεραιότητες σε ό,τι αφορά την οικονομία, σε ό,τι αφορά την αγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανεφέρθηκα ήδη στις τρεις προτεραιότητες απασχόληση, επιχειρηματικότητα και επιχειρήσεις. Το 2016 η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων θα συνεχίσει να λειτουργεί, να αναπτύσσεται και είχαμε δεσμεύσει, πιστώσεις, αλλά θα έχουμε λήψει το 2016. Είναι λοιπόν επιτακτική ανάγκη να συνεχίσει να είναι λειτουργικό το πρόγραμμα αυτό και προφανώς χρειάζεται επαρκής χρηματοδότηση προκειμένου να ανταπεξέλθουμε στο ύψος των δεσμεύσεων Και προφανώς θα πρέπει αυτά να α, χορηγηθούν ως αναλήψεις υποχρεώσεων. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει ανάληψη των ευθυνών. Και προφανώς θα το θεωρήσουμε αν υπάρξουν προβλήματα ε, σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση προγραμμάτων όπως το Connecting Europe. Όταν εγκρίναμε το EFCI το πρόγραμμα Juncker, δεσμευθήκαμε. Δεσμευθήκαμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να περιορίσουμε στο βαθμό του δυνατού τον αντίκτυπο στον ορίζοντα 2020 και στο Connecting Europe. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν έκανε μια πρόταση. Παρ' όλα αυτά το Συμβούλιο επέδειξε μια στάση η οποία μόνο ως πρόκληση προς το Κοινοβούλιο μπορεί να θεωρηθεί. Γιατί περικόπτουν τα προγράμματα αυτά, περικόπτουν τον ορίζοντα 2020, περικόπτουν την ε, διευκόλυνση Connecting Europe και συνοπτικά, για να κάνω μια ανακεφαλαίωση, πρέπει να σας πω ότι το Κορεπέρε ενέκρινε μια θέση η οποία περιλαμβάνει μείωση των ε, να δεσμεύσουμε 543 εκατομμύρια στις πληρωμές 1,4 δισεκατομμύρια περικοπές. Και αυτές οι περικοπές είναι σε σχέση με το σχέδιο προπολογισμού που έχει καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτό ήδη ήταν μειωμένο σε σχέση με αυτά που προβλέπονται στο πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτό ομόφωνα εγκρίθηκε από την Κορεπέρ. Περικοπή λοιπόν. Περικοπή περικοπή επί ενός προϋπολογισμού που ήταν ήδη μειωμένος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ύστερα στο τμήμα 1α Έχουμε 73 εκατομμύρια για τον ορίζοντα 2020 και 205 περικοπές στις πληρωμές και περικοπές επίσης στο Connecting Europe Facility. 16,3 και 10,7 αντίστοιχα στις δεσμεύσεις και στις πληρωμές. Σε αναλήψεις υποχρεώσεων και στις ε, πληρωμές. Περικοπές οι οποίες τελικά θα καταλήξουν να κλείσουν προγράμματα στο 2α και στο 3. Τα προγράμματα ευελιξίας, για παράδειγμα, 124 εκατομμύρια ευρώ που προορίζονται και στην αντιμετώπιση του θέματος των μεταναστών και των προσφύγων. Το Συμβούλιο δεν έχει περικόψει κάποια προγράμματα για το άσυλο και τη μετανάστευση, ούτε έχει περικόψει χρηματοδότηση για την ιστορική ασφάλεια. Ωστόσο, ωστόσο, έχει μειώσει σοβαρά το ποσό που σκοπεύει να χορηγήσει στα εργαλεία ευελιξίλια. Στην ε, τμήμα 4, 163 ε, εκατομμύρια και 450 ε, εκατομμύρια στις αναλήψεις υποχρεώσεων και στις πληρωμές. Αντίστοιχα, μιλάμε για σοβαρές περικοπές που φυσικά θα έχουν αντίκτυπο στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Όλες αυτές οι περικοπές λοιπόν είναι απαράδεκτες και για τις ε, εξωτερικούς οργανισμούς, ε, περικοπή στις αναλήψεις υποχρεώσεων, λίγο πολύ για όλες τις εξωτερικές υπηρεσίες. Όλα αυτά τα θεωρούμε απαράδεκτα. Και το προχωράει ακόμα το επιχείρημα, το Συμβούλιο. Δηλώνει ότι, λέγοντας ότι κάνει περικοπές όπου υπάρχει μικρότερη απορρόφηση των πόρων. και λιγότερη εφαρμογή, δηλαδή δεν υπάρχει ε, ικανότητα απορρόφησης και εκτέλεσης των προγραμμάτων. Ομολογμένως υπάρχουν προγράμματα τα οποία είναι εξαιρετικά, αλλά υπόκειται περικοπές στο 1α και στο 3, το Connecting Europe, το Europe for Citizens, στον τμήμα 4 προγράμματα τα οποία έχω ήδη αναφέρει προγράμματα πρόληψης ε, συγκρούσεων για τη μείωση της φτώχειας ε, στην Μεσόγειο. Όλα αυτά λοιπόν πετσοκόβονται. Και το Κοινοβούλιο έχει σαφή εντολή, την οποία την ενέκρινε με μεγάλη πλειοψηφία. Άρα, τη στάση του να την εκτιμήσουμε ως απαράδεκτη. Και ως εκ τούτου, θα προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία ευελιξίας που θα μας επιτρέψουν να χρησιμοποιήσουμε τα περιθώρια που έχουμε και να αυξήσουμε τις ε, πληρωμές. Και αντιστοίχως θα επιδείξουμε και υπευθυνότητα. Είμαστε φιλόδοξοι και στεναροί. Και σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να ζητήσουμε από το Κοινοβουλίο να ανταπεξέλθει και να, τα, να έρθει στο ύψο των περιστάσεων σε ό,τι αφορά τι αναλήψει υποχρεώσεων. Και εδώ θα ήθελα να τονίσω τον παράγοντα τη μετανάστευση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αξίε όπω η αλληλεγγύη, ο σεβασμό τη ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Πρόκειται για αναπαλατρίωτε αξίε. Και γι' αυτό λοιπόν είναι απαράδεκτο το Συμβούλιο να λέει ότι από πλευρά προπολογισμού, Α, κοιτάξτε, δεν θέλουμε να κάνουμε τίποτα, θέλουμε περικοπέ. Εντάξει, να μιλάμε εμένα, αλλά να μην κάνουμε τίποτα. Και οι πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση στρέφονται προ την πλευρά των τριών θεσμικών οργάνων, κατηγορούν και επιρρύπτουν ευθύνε στην Ευρώπη. Εδώ το Κοινοβούλιο λοιπόν πρέπει να επιδείξει ότι μπορεί να προασπιστεί τις αξίες της και τις προτεραιότητές της και μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της μετανάστευσης. Ευχαριστώ κύριε Γενική Εισηγητή. Χαίρομαι που βλέπω να έχετε επιστρέψει όλοι από τις δεκοπές ε, σε φόρμα. Τα πρώτα σώπα σας εκτενοβολούν. Είστε όλοι ξεκούραστοι. Πιστεύω ότι η επιστροφή θα είναι ιδιαίτερα ζωντανή. Και σε δημοσιονομικά θέματα σκοπεύουμε να ακουστεί η φωνή μας. Ευχαριστούμε Μανουέλ για αυτή την παρουσίαση. Καλό τώρα τον κύριο Ντεπρέ να μας γνωρίσει τις παρατηρήσεις του για τα υπόλοιπα τμήματα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σχετικά σύντομος στην παρούσα διότι ήδη έχουμε επιτύχει την έγκριση στην Ολομέλεια του Προεπιλογισμού του Κοινοβουλίου. Υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα όμως το πώς θα αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες, τις δημοσιονομικές συνέπειες για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για το οργανόγραμμα από την αναγνώριση μιας νέας πολιτικής ομάδας. Θα σας μιλήσω για αυτό σε λίγο. Διότι πρέπει να περιμένουμε να αποφασίσει το Προεδρείο του Κοινοβουλίου για τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα σε γενικές γραμμές ω στάση ε, και δεδομένου το Συμβούλιο έκανε σημαντικές ε, περικοπές τυφλά εδώ παντού ε, επιθυμώ να αποκαταστήσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με δύο εξαιρέσεις. Η πρώτη αφορά το δικαστήριο. Θεωρώ ότι όταν συμφωνεί κάποιος για μια αύξηση για το δικαστήριο πρέπει να λάβει σοβαρά οτιδήποτε συνέπειε θα έχει αυτό σε θέματα οργανογράμματο και σε χρηματοοικονομικά θέματα. Για αυτό το σημείο λοιπόν θα ζητήσω από την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο να πάνε λίγο πιο πέρα από αυτά που πρότεινε η Κομισιόν, διότι θεωρώ ότι είναι απαραίτητο, είναι δικαιολογημένο και θα ήταν ανεύθυνο να μην γίνει. Για τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα, σε γενικέ γραμμέ όπω είπα, ε, μιλάμε για επιστροφή στο σχέδιο προπολογισμού της Κομισιόν με μια ή διορθώσεις που θα σας αναφέρω αργότερα. Αυτό σχετίζεται με τη συζήτηση που θα κάνουμε σε σχέση με τις γενικές ε, κατευθύνσεις που θα προσθέσει ο συνάδελφος κ. Φερνάνδες για τον προπολογισμό της Κομισιόν. Αυτά κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Αυτά επιθυμούσα να πω στην παρουσία Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ντεπρέ. Το λόγο έχουν τώρα οι σκιώδεις και οι λοιποί συνάδελφοι. Έχω τον κύριο Μάνκα στην ε, λίστα μιλητών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Έχω δύο σχόλια. Το πρώτο αφορά την εκθέση του κ. Φερνάνδες ε, υποστηρίζω τα όσα μας είπε και πραγματικά πρέπει να αναφέρουμε την ανοργανωσιά και τις χαοτικές αποφάσεις του Συμβουλίου ειδικότερα στο θέμα της μετανάστευσης. Αν δεν θυμάστε, στο προπολογισμό της Frontex εδώ και χρόνια ζητάμε αύξηση του προπολογισμού του Frontex και τελικά όταν τα πράγματα πραγματικά δυσκολεύουν ξαφνικά το Συμβούλιο συμφωνεί σε, σε τριπλασιασμό του προπολογισμού. Το ίδιο αφορά και ορισμένε άλλε προτεραιότητε. Ορισμένε προτεραιότητε προέρχονται μένα από το Συμβούλιο, αλλά αυτό δεν προβλέπει προπολογισμό για αυτέ. Εγώ ήμουν εισηγητή και για τα άλλα θεσμικά όργανα, οπότε μπορώ να σα αναφέρω δύο λόγια. Πρόκειται να συζητήσουμε το απόγευμα με το Γενικό Γραμματέα, τον προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οπότε δεν θα τον αναφέρω τώρα. Αλλά όσον αφορά τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα, το Συμβουλίο ε, επαναλαμβάνει τον προπολογισμό και ορίζει τον προπολογισμό για ορισμένα θεσμικά όργανα χωρίς κανείς να γνωρίζει γιατί έγιναν ορισμένες περικοπές. Πιστεύω ότι θα πρέπει να επιστρέψουμε τον προπολογισμό αυτών των θεσμικών οργάνων και να ζητήσουμε από το Συμβουλίο να μας δώσει εξηγήσει. εξηγήσεις για αυτές τις περικοπές. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Επόμενος συναδέλφος, η κυρία Μούδη. Thank uh, Ευχαριστώ για να απαντήσω στο Γενικό Εισηγητή και να υπερθεματισώ και τα όσα είπε για τις δύο προτεραιότητες ε, που έχουν ιδιοριστεί για τον προπολισμό του 2016 όσον αφορά την ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα της μικρομεσαίας επιχειρήσης. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι ο προπολογισμό του ορίζοντα 2020 πρέπει οπωσδήποτε να ενδυναμωθεί. Μαζί με αυτό έχουμε και το ότι πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό που κάνουμε καλύτερα ως Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι κυρίως η ανάπτυξη και ιδιαίτερα μέσω του Horizon 2020. Αλλά αυτό που λέμε και κατά επανάληψη εδώ, ε, η σημασία πρέπει να δοθεί στο ζήτημα της μετανάστευσης και στην ε, κρίση ε, των προσφύγων που αντιμετωπίζουμε τώρα πρέπει οπωσδήποτε να διατηρήσουμε τη δημοσιονομική ευθύνη, αλλά αυτό που θα κάνουμε συλλογικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να γίνει βάση αυτών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κυρία Κελμά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τους συζητητές και τους σκιώδες. Συμφωνώ ε, και έχει δίκαιο ο κύριος Φερνάντες σε πολλά από όσα είπε. Χρειάζεται περισσότερη ειλικρίνη εδώ και εντιμότητα και στον προϋπολογισμό. Δηλαδή, τα κράτη-μέλη δεν μπορούν από τη μια να λέγουν ότι θέλουν τον ουρανό με τα άστρα, αλλά μετά δεν θέλουν να το χρηματοδοτήσουν αυτό. Από την άλλη όμως θα πρέπει να προσέχουμε και το εξής τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να χρηματοδοτούν τον προϋπολογισμό και πρέπει να βρούμε μια ισορροπία. Άμεσα σε αυτά που επιθυμούν να χρηματοδοτήσουν τα κράτη-μέλη και το τι ε, επιθυμητό αποτέλεσμα θα προκύψει. Πολλά σωστά υπόθηκαν και πολλοί τομεί. Θέλω όμω να προειδοποιήσω για κάτι. Να μην αφήσουμε να δημιουργηθεί εντύπωση ότι όπου υπάρχουν προβλήματα στην οικονομία, θα πρέπει να κληθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει και θα χρηματοδοτήσουμε το πρόγραμμα αυτό και θα πάνε όλα καλά. Δεν ισχύει αυτό, διότι όχι απλώς δεν υπάρχουν χρήματα για να το χρηματοδοτήσουν, αλλά είναι και πολύ λανθασμένος ο δρόμος αυτός, να τον ακολουθούμε. Δηλαδή, ο ακτιβισμός δεν είναι στρατηγική. Για ποιο λόγο, λοιπόν, χρειαζόμαστε περισσότερη ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα και πώς επιτυχάνεται αυτή. Δεν γίνεται με επιδοτήσεις. Εμείς ένα σωρό προγράμματα ε, εφευρίσκουμε και προσπαθούμε να επιδοτούνται αυτά όσο γίνεται περισσότερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν οδηγεί από μόνο του σε μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Εμεί θα πρέπει να δούμε πού μπορούμε να θέσουμε κέντρα βάρου, να επικεντρωθούμε και να περιοριστούμε σε συγκεκριμένα πράγματα και να δίνουμε κίνητρα ε, έτσι ώστε να αναπτυχθεί μια διαδικασία που να αποκτήσει ίδια δυναμική και πορεία. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για τις συζητήσεις που κάνουμε για τον προπολογισμό. Ιδιαίτερα δε σε αυτή την τραγωδία με τους πρόσφυγες και τα δράματα που βλέπουμε να εκτελήσονται και ε, σε ό,τι αφορά τη μεγάλη αυτή ε, προσέλευση, το κύμα προσφύγων προς την Ευρώπη. Εδώ πρέπει να δράσουμε και θα ήμουν ε, απολύτως πρόθυμος και αμέσως να υπερψηφίσω περισσότερα κονδύλια, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και μια συνολική θεώρηση και πρόγραμμα για τους πρόσφυγες. Αυτό μέχρι τώρα δεν υπάρχει. Βέβαια θα πρέπει πρώτα να ανακουφιστεί η επίγουσα κατάσταση, τα, τα δεινά αυτών των ανθρώπων. Αλλά εάν θέλουμε να δαπανίσουμε ευρωπαϊκά κονδύλια χρειάζεται και ευρωπαϊκό σχέδιο, το οποίο στερούμαστε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ας εκπονήσουμε αυτό το σχέδιο και δεσμευτικά να καθορίσουμε τι θα ισχύει. Γιατί διαπιστώνω ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή, κατά την άποψή μου πάντα, κινδυνεύει να χάσει ε, τη φήμη της όλοι ξέρετε ότι η συνθήκη του Μαστρίχ δεν αξίζει καν ούτε το χαρτί στο οποίο είναι γραμμένη. Υπάρχει και η περίφημη συνθήκη, η σύμβαση του Δουβλίνου που στο μεταξύ έχει γίνει και αυτή κουρελόχαρτο να μην κάνουμε πολιτικές βιτρίνες με διάφορες συνθήκες και συμβάσεις που τελικά δεν τηρούνται. Σίγουρα αυτό δεν το περιμένουν από εμά οι πολίτες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βάλη. Ναι, ευχαριστώ. ευχαριστώ τους δύο συγγητές. Ήθελα απλά να κάνω μια-δυο διευκρινήσεις και παρατηρήσεις όσον αφορά το κομμάτι που αφορά τα υπόλοιπα τμήματα. Φυσικά το Συμβουλίο δεν άγγιξε τον προπολογισμό του Κοινοβουλίου ε, δύναμη αυτής της ε, απόφασης. Ε, είναι παράλογο να διατηρούμε προνόμια μεταξύ των ε, θεσμικών οργάνων θέλουμε εμείς να προσπαθήσουμε να περιοριστεί η υπερβολική σπατάλη χρημάτων οι άλλες περικοπές είναι μικρές παρότι ε, αρκετά σημαντικές θέλω να σταθώ σε δύο περιπτώσεις στην ε, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών. Σίγουρα στο παρελθόν έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εκπροσώπηση στις Βρυξέλλες επιχειρήσεων, εργαζομένων αλλά έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα θεσμικά όργανα και τα νομοθετικό σύστημα έχουν χάσει την χρησιμότητά τους. Εμείς προτείνουμε τροπολογίες σημαντικές ε, για αυτούς τους οργανισμούς με περικοπές του 20% για σημαντικά κονδύλια. Πρέπει να κλείσουν ε, ή να αναδιαργωνωθούν αυτά τα δύο όργανα, αλλά δεν μπορούμε να σπαταλάμε πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Τώρα, όσον αφορά τη μείωση του προσωπικού κατά 5%, συμφωνούμε απόλυτα. Αλλά θα θέλαμε να γίνει και μια πιο σημαντική συζήτηση που θα αφορά όχι μόνο τον αριθμό αλλά και το ύψος της αμοιβή του. Αυτό είναι ένα θέμα που εμείς προσπαθούμε να προωθήσουμε και στον έλεγχο του προπολογισμού, διότι πήγα να δω τους πίνακες ε, αμοιβών των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μου φαίνονται δυσανάλογα υψηλές σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα. Τα οργανογράμματα ε, έχουν ε, πολλά νούμερα για διάφορους βαθμούς ε, αντίθετα από ό,τι γίνεται σε φυσιολογικές επιχειρήσεις ή οργανισμούς. Πολλοί κόσμος έχει αρκετά υψηλού μισθού Ε, επ' αυτών των σημείων θα επικεντρωθούν οι τροπολογίε μα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Επόμενος ομιλητής, ο κ. Χριστοφόρου. Ε, πιστεύω ότι είναι ατυχής η, η πολιτική που εφαρμόζει το Συμβούλιο όσον αφορά την προσέγγιση του προπολογισμού και θα συμφωνήσω πλήρως με τον αγαπητό συνάδελφο τον κύριο Φερνάντες εφόλης της ύλης, δηλαδή ότι αυτή η πολιτική είναι αντιφατική γιατί εάν αντιπαραθέσουμε εδώ τις δηλώσεις, τις θεωρητικές δηλώσεις που κάνει το Συμβούλιο για τον προϋπολογισμό και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δηλώσεις πλειοδοτικές που ουσιαστικά θέλουν και άλλα χρήματα και στην πράξη έρχονται να μειώσουν αυτά τα οποία ουσιαστικά οι ίδιοι ζητούν καθημερινά μέσα από τις δικές τους δηλώσεις. Όμως θεωρώ ότι εάν το Ευρωκοινοβούλιο περάσει αυτόν τον προϋπολογισμό με αυτήν την πολιτική, ουσιαστικά και το Ευρωκοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βρεθεί αντιφατική με τον ίδιο της τον εαυτό και με την ίδια της την πολιτική. Δηλαδή, Εμεί ω Ευρωκοινοβούλιο στηρίξαμε και υποστηρίξαμε ότι για να αντιμετωπιστεί ο αποπληθωρισμό που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να ρίξει χρήματα στην αγορά 3 εκατομμύρια. Την ίδια στιγμή εμεί που υποστηρίζουμε να καταπολεμήσουμε τον αποπληθωρισμό και να δώσουμε χρήματα για την ανάπτυξη, ουσιαστικά αποδεχόμαστε έναν προπολογισμό που κινείται στην εντελώ αντίθετη κατεύθυνση. Να στερήσει χρήματα για την ανάπτυξη, να ενισχύσει περαιτέρω τον αποπληθωρισμό και ουσιαστικά να φαντάζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο έχει αντιφροτική πολιτική, αλλά δεν είχε καθόλου πολιτική και όλα αυτά τα ζητήματα. Δυστυχώ θα βρεθούμε για μια ακόμη φορά να απαξιώνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν ξέρει τι θέλει και δεν ξέρει τι τη γίνεται, γιατί η πολιτική του προπολογισμού τη θα είναι σε πλήρη σύγκρουση με τι εξαγγελόμενε πολιτικέ για ανάπτυξη, για αλληλεγγύη, η αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, η αντιμετώπιση της ανεργίας, για στήριξη προγραμμάτων που έχουν να κάνουν με την έρευνα και την καινοτομία, ουσιαστικά ακυρωνόμαστε. Και ως Ευρωκοινοβούλιο ακυρωνόμαστε. Δεν έχουμε θέση σε αυτήν την πολιτική. Τελικά πρέπει να μας προβληματίσει. Άλλη πολιτική έχει το Συμβούλιο, άλλη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, άλλη το Ευρωκοινοβούλιο πολλές φορές. Είναι ευτυχές το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμπίπτει με το Ευρωκοινοβούλιο. Δεν μπορεί λοιπόν το Συμβούλιο ως όργανο να ακυρώσει και τον εαυτό του και την ευρωπαϊκή πολιτική και την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δηλαδή είναι θέμα αρχή. Εκεί πρέπει να σταθούμε. Σίγουρα δεν θα βρεθεί τρόπο εκ μέρου του να δικαιολογήσουν τι μειώσει, όμω εγώ είμαι εξ εκείνων που πιστεύω αν θέλουν να κάνουν μειώσει υπάρχουν περιττέ δαπάνε ή σπατάλε που μπορούν να τι περιορίσουν. Μπορούν να περιορίσουν τη γραφειοκρατία και επειδή έγινε και μια αναφορά για το Ευρωκοινοβούλιο, εδώ αντί να δούμε τα μεγάλα ζητήματα, που είναι αυτά που είναι οι περικοπές, κάποιοι από εμάς αρχίζουμε να αυτοπυροβολούμαστε. Δηλαδή αντί ο στόχος ολονών να είναι να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε την εσφαρμένη πολιτική του Συμβουλίου, αρχίσαμε πάλι το παραμύθι του Ευρωκοινοβούλιο έχει σπατάλες. Καλά, το Ευρωκοινοβούλιο είναι το 1% ή το 2% του προπολογισμού. Ε, κάποιοι αν είναι τόσο τολμηροί, γιατί δεν καταπιάνονται με τα αγροτικά προγράμματα που είναι το 40%. Είναι πολύ πιο εύκολο να περιορίσει δαπάνε ή σπατάλε από έναν κομμάτι που λέγεται ω παράδειγμα το φέρω. Δεν λέω ότι πρέπει να πάμε να κόψουμε από την αγροτική οικονομία. Αλλά εάν κάποιοι είναι τόσο ευαίσθητοι για σπατάλε, πιο εύκολα θα βρει σπατάλε εκεί που διαθέτει το μισό σου προπολογισμό από εκεί που διαθέτει το 1 με το 2%. Και επειδή είναι ιδιαίτερα λαϊκιστικό το ζήτημα, από μόνοι μας θα στρέψουμε την προσοχή σε κάτι ανύπαρκτον, μη σημαντικό και ουσιώδες για να το παίξουμε υπεράνω και θα χάσουμε την ουσία και την μεγάλη εικόνα που είναι να στηρίξουμε αυτά που είπε ο αγαπητός συνάδελφος ο Τζοζέ, την ουσιαστική πολιτική. Γι' αυτό για μένα ουσιαστική πολιτική είναι να βασιστούμε σε αυτά ως στρατηγική που ανάφερε ο Φερνάντης προηγουμένως, να διεκδικήσουμε από το Συμβούλιο και πιστεύω ότι αυτός ο προϋπολογισμός δεν θα είναι ούτε αναπτυξιακός αν περάσει ως έχει και πρέπει να το πούμε ούτε αναπτυξιακός ούτε προπολογισμό αλληλεγγύη, ούτε προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά. Θα είναι ένα προπολογισμό που το Συμβούλιο εν διαγνία του πολλέ φορέ ή ακόμα και παρασυρώμενο πήγε και έκανε αυτέ τι οριζόντιε περικοπέ. Άρα πιστεύω να μείνουμε στα μεγάλα, στα σημαντικά, να μην χάσουμε το δάσο για χάρη του δέντου. Ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τόμας. Oui, merci, Monsieur le Président. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον εισηγητή και να πω ότι συμμερίζομαι την ανάλυση, συμφωνώ με την ανάλυση αυτή και μπορούμε να υποστηρίξουμε ε, τα όσα ακούσαμε. Θα μιλήσω λίγο σκληρά, λίγο ομά ίσως, που ουσιαστικά θα μοιάζουν με αυτά που μόλις ακούσαμε. Βρισκόμαστε ενώπιον ενός συμβουλίου ε, που δεν έχει λογική. Ε, ζητά όλο και περισσότερα ευρωπαϊκά μέσα από τη μία. Αφετέρου θέλει να συμβάλλει όλο και λιγότερο και έτσι ξαφνικά κάνει διάφορες ανακοινώσεις ε, για τους μετανάστες, ε, για την ανάπτυξη, ε, για τους πρόσφυγες, για την υποστήριξη της ανάπτυξης και τελικά πάει και επιλέγει περικοπές δημοσιονομικές που έρχονται σε αντίθεση με τις ανακοινώσεις που κάνει. Έτσι λοιπόν δεν μπορεί να κρατήσει τις υποσχέσεις του. Οι διαπραγματεύσεις ήταν πάρα πολύ δύσκολες στο πλαίσιο του πολιτού δημοσιονομικού πλαίσιου, εξαιρετικά δύσκολες. Και εμείς ελπίζαμε ότι θα είχαν ε, σεβαστεί και τα δύο μέρη το συμβιβασμό που επιτεύχθη, αλλά δεν συνέβη αυτό και το είπε και ο κύριος Φερνάνδες. Κάθε χρόνο έχουμε περικόπες του προπολογισμού σε σχέση με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, χωρίς να μιλήσουμε για τα προβλήματα πληρωμών ε, που έχουν συζητηθεί εκτενώς σε αυτήν εδώ την Επιτροπή. Δεν έχει λοιπόν συνοχή, δεν κρατάει το λόγο του, περιφρονεί το κοινοβούλιο παρότι είμαστε τη δημοκρατία και κυρίως δείχνει ανευθυνότητα. Διότι ε, τι, ε, αναμένουν οι πολίτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση να τους βγάλει από την αδυναμία, από την ακινησία, να μπορέσει να τους καταστήσει χρήσιμους, ε, να χρησιμεύσουμε εμείς. Πώς θα το κάνουμε αυτό χωρίς τον απαραίτητο προπολογισμό. Ξέρετε, τα κράτη-μέλη δεν επιλέγουν κάθε χρόνο τη συμμετοχή τους. Η συμμετοχή των κρατών μελών δεν είναι ότι κάθε χρόνο βάζει ο καθένα ό,τι θέλει. Υπάρχουν ποσοστά. Ανάλογα με το ακαθάριστο προϊόν, το οποίο ε, δεν είναι συζητήσιμο, ούτε διαπραγματεύσιμο. Παρότι το συζητάμε μερικέ φορές. Ίσως αυτό θα έπρεπε να το ξαναδούμε. Και πολλές φορές ακούμε το ευρωπαϊκό έργο, δεν το, συμφωνούν όλοι με αυτό, ακούμε πολλές επικρίσεις, αλλά όπως και να το κάνουμε υπάρχουν μερικά θέματα στα οποία συμφωνούμε. Συζητήσαμε για τις επενδύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Το κοινοβούλιο αυτό ε, με πολύ μεγάλη πλειοψηφία υποστήριξε αυτή την ε, επένδυση για την ανάπτυξη και την απασχόληση Είχαμε τεράστιες πλειοψηφίες εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το ίδιο και για τους πρόσφυγες. Ε, ξέρετε, εντός του κοινοβουλίου αυτού είχαμε μια συντριπτική πλειοψηφία ε, υπέρ αυτών των ζητημάτων. Όλα αυτά για να πω ότι εδώ και αρκετά χρόνια έχουμε μια σημαντική ασυνεννοησία μεταξύ των προσδοκιών των Ευρωπαίων ε, των ε, σχετικών ανακοινώσεων αφενός και των ε, προπολογισμών που εγκρίνονται. Το Κοινοβούλιο δεν ευθύνεται για αυτή τη διαφορά απόψεων. Η αντιπαράθεση τώρα με το Συμβούλιο θα γίνει πιο ορατή, διότι, ξέρετε, μέχρι στιγμής θεωρούσαμε ότι όλοι είμαστε μέσα στο στον ίδιο κουβά, ξέρετε, το στο ίδιο τσουβάλιο το, η Κομισιόν, το Κοινοβούλιο και ε, το Συμβούλιο, αλλά αυτό πρέπει να το τονίσουμε ότι δεν είναι πια έτσι, ώστε να το δουν και οι πολίτες μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Συναδέλφοι, έχουμε καθυστερήσει λίγο σε σχέση με το πρόγραμμα. Θα ήθελα λοιπόν οι υπόλοιποι ομιλητές να περιοριστούν στα δύο λεπτά, αν είναι δυνατόν. Παρακαλώ, κύριε Σαλή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Το σχέδιο προπολογισμού που προτάθηκε από την Κομισιόν εστιάστηκε σε προτεραιότητες. Οι προτεραιότητες αυτές είχαν οριστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν θα μπω τώρα σε λεπτομέρειες εδώ, αλλά πιστεύω ότι η έκθεση του κυρίου Φερνάντες ε, τα, περι... τα συμπεριέλαβε όλα. Ε, πρέπει να πω ότι εμείς υποστηρίζουμε τις πολιτικές που αναφέρει. Όλες οι προτεραιότητες που αναφέρθηκαν από τον κύριο Φερνάντες και από τους λοιπούς συναδέλφους, όπως η Ενεργειακή Ένωση, η Απασχόληση, η Δημιουργία Θέσεων Εργασίας, όλες αυτές οι προτεραιότητες αποσκοπούν στο να δώσουν μια απάντηση στα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, στις νέες εξελίξεις. Ωστόσο, βλέπουμε ξαφνικά μια περικοπή στον προπολογισμό αυτό της τάξης του 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αν το συγκρίνουμε με τον προηγούμενο προπολογισμό, πρόκειται για μια... Μας λένε ότι είναι αύξηση ουσιαστικά, αλλά αν υπολογίσουμε τον ε, πληθωρισμό, πρόκειται για περικοπή και αυτό θα έχει πολύ αρνητικές συνέπειες. Αν ε, συζητήσουμε λεπτομερώς όλες τις περικοπές θα δούμε ότι στις, ε, ε, στους τίτλους 1, στις 1 1α, 1β, 2 και 4 η μεγαλύτερη περικοπή βρίσκεται υπό την επικεφαλίδα 4 Global Europe. Μιλάμε για περικοπή σχεδόν του, του 5%. ουσιαστικά το Συμβούλιο προτείνει πολλές περικοπές, όπως είπα. Οι περικοπές αυτές θα δημιουργήσουν προβλήματα. Είναι σαφές ότι οι περικοπές αυτές αφορούν τομείς προτεραιότητας που έχουν ήδη συμφωνηθεί μεταξύ Συμβουλίου, Επιτροπής και Κοινοβουλίου. Οι περικοπές υπό την επικεφαλίδα 4 θα θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο τις πολιτικές, ε, ε τις μεταναστευτικές πολιτικές μας και ε, βλέπετε τι γίνεται τους τελευταίους μήνες η μετανάστευση αρχίζει να αποτελεί επίγον πρόβλημα και ε, πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε μια λύση. Ωστόσο, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω μετά από όλες αυτές τις περικοπές ειδικότερα στο μέσο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας πώς θα αντεπεξέλθουμε στην εισρωή, στο κύμα αυτό προσφύγων και μεταναστών. Είναι σοβαρό πρόβλημα. Δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε. Πιστεύω ότι η θέση μας θα πρέπει να διακατέχεται από συνοχή και πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια να επιτύχουμε καλά αποτελέσματα στον επόμενο τριμερή διάλογο ενωμένοι όσον αφορά την προσέγγιση μας, τη διαπραγματευτική μας προσέγγιση με το Συμβούλιο και να παραμείνουμε πιστοί στα όσα είπαν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Ο κύριος Τζάνι. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα είμαι σύντομο. Ήθελα να απαντήσω στον συνάδελφο του ΕΛΚ για τις περικοπές και τις πατάλες. Ίσως γι' αυτό να υπάρχουν ε, ε, σπατάλες ε, δεύτερης κατηγορίας. Ξέρετε, καθήκον μας είναι να βλέπουμε τις σπατάλες και του ενός ευρώ ε, και το 1 ευρώ των πολιτών μα που σπαταλάτε δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Αυτή είναι η προσέγγιση που έχουμε χρησιμοποιήσει εμεί. και αν είναι να περικόψουμε μη παραγωγικέ ε, δαπάνε για τη λειτουργία του Κοινοβουλίου, ακόμη και αν αυτό αντιστοιχεί στο 1% του προπολογισμού τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστεύω ότι αποτελεί καθήκον μα να τι βρούμε, να τι εντοπίσουμε και να τι διαγράψουμε. Δεν υπάρχουν για μένα ε, σπατάλες, επαναλαμβάνω, κατηγορία Α και Β. Υπάρχουν απλά σπατάλε δημόσιου χρήματο. Γενικότερα όσον αφορά τον προϋπολογισμό, έχω ήδη εκφράσει τη θέση μου στους συναδέλφους προηγουμένως στη συνεδρίαση των συντονιστών, αλλά υπάρχουν ένα-δύο σημεία τα οποία θα ήθελα να επισημάνω. Το πρώτο αφορά την απόλυτη ασυνοχή του Συμβουλίου όσον αφορά τις θέσεις του πιστεύω ότι πρέπει να περιγράφει πιο καθαρά τι προτεραιότητε του να, για να μπορούμε να καταλάβουμε προ τα πού θέλει να πάει, ποιο είναι το όραμα του Ευρωπαϊκού προπολογισμού σύμφωνα με το Συμβούλιο. Για παράδειγμα, παρατηρούμε ορισμένα κονδύλια στον προπολογισμό όπου το Συμβουλίο έχει προβεί σε περικοπές 20, 30, 40% τόσο για αναλήψη υποχρεώσεων όσο και για πληρωμές. Τι σημαίνει αυτό αν δούμε πέρα από τα νούμερα. Σημαίνει ότι το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη δεν πιστεύουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, στο συγκεκριμένο κονδύλιο. Οπότε εκεί πρέπει να σκεφτούμε, να συζητήσουμε μαζί με το Συμβούλιο. Αν δεν πιστεύετε αυτή τη γραμμή του προπολογισμού, αυτό το κονδύλιο, έχει νόημα να συνεχίσουμε να τη χρηματοδοτούμε ή όχι. Αυτό το δίλημα πρέπει να επιλύσουμε. Εάν πιστεύουμε, συνεχίζεται επαρκή χρηματοδότηση. Αν όχι, ε, δεν υπάρχει λόγο να ρίχνουμε άλλα χρήματα εκεί, απλά για να υπάρχει. Όσον αφορά τι πληρωμέ και εδώ η θέση του Συμβουλίου είναι εντελώ αντιδιαμετρική. Εμείς ε, συνεργαζόμαστε με την Επίτροπο Γεωργίευα για να επιλύσουμε το πρόβλημα των πληρωμών, των ε, ε, ανεξόφλητων τιμολογίων. Γίνεται τεράστιε προσπάθειε και ξαφνικά το Συμβούλιο έρχεται και μας κάνει μια πρόταση αύξηση αυτής της διαφοράς μεταξύ αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών. Πρέπει να το καλύψουμε αυτό το χάσμα. Υπάρχουν δύο τρόποι. Είτε να μειώσουμε τις, ε, δεσμε... Ε, τις αναλήψεις υποχρεώσεων, είτε να αυξήσουμε τις πληρωμές. Εγώ είμαι για το ε, πρώτο, αλλά το Συμβούλιο πρέπει να αποφασίσει. Τώρα για το τμήμα 4, όπως είπε ο συνάδελφος του Άλντε. Ναι, και αυτό είναι ένα μέσο επίλυσης του προβλήματος των μεταναστευτικών ροών να εφαρμόσουμε μια ικανοποιητική πολιτική βοήθειας παρέχοντας κονδυλία στα διαφορετικά κράτη, ίσως θα δημιουργήσουμε τις συνθήκες για να υπάρχουν συνθήκες τέτοιες στις χώρες καταγωγής ώστε να μην υποχρεούνται οι άνθρωποι να μεταναστεύουν. Και εδώ λέμε να δίνουμε χρήματα, αλλά την άλλη τα κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι ο πρώτος εξαγωγιάς όπλων σε αυτές τις ε, περιοχές σειράξεων, εκμεταλλεύεται τους πόρους των χωρών αυτών. Δηλαδή από τη μία δίνουμε λεφτά και από την άλλη δημιουργούμε τις συνθήκες με τις οποίες ε, οδηγούνται αυτοί οι άνθρωποι λόγω πολέμου να έρθουν σε εμά. Και εκεί χρειάζεται λιγάκι πιο συνεκτική προσέγγιση από του Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Τελευταία Τελευταίο είναι κατάλογο Μιλτών. κύριε Μερικάλη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Λοιπόν, δεν είναι δύσκολο να συμφωνήσεις με τις αρχικές θέσεις του κυρίου Φερνάντες και με τις επικρίσεις που ακούμε για το Συμβούλιο επανειλημμένα. Δεν χρειάζεται να προσθέσω τίποτα, έχω καλυφθεί απολύτως. Θα ήθελα μόνο να τονίσω ένα σημείο. Αν θέλετε, πώς να το πω, κάτι που έχει ευθύνη και το Κοινοβούλιο σε αυτό. Εμείς δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από την αδιαλαξία του Συμβουλίου για να τελειώσουμε στο παραπέντε ή στο παραένα ε, υποπίεση τη διαπραγμάτευση και τελικά να περιορίσουμε όσο γίνεται την αδιαλαξία. Υπάρχει και πολιτική ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του, του Κοινοβουλίου. Εδώ και στο Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε ένα μεγάλο συνασπισμό των δύο μεγάλων πολιτικών ομάδων που φέρουν ευθύνη και ρητή για όλες τις πολιτικές και δεν μπορούμε απλώς έτσι να ξεφεύγουμε απορρίπτοντας το Συμβούλιο και να τα ρίχνουμε όλα στην αδιαλαξία των κρατών μελών. Έχει έρθει η ώρα της πολιτικής και μάλιστα της ευρωπαϊκής και συνολικής πολιτικής. Δεν μπορούμε να συζητούμε πώς θα περιορίσουμε ή θα λαχιστοποιήσουμε τις περικοπές του Συμβουλίου. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι αν θα διπλασιάσουμε, να τριπλασιάσουμε ή να τετραπλασιάσουμε ε, τα κονδύλια για τους πρόσφυγες. Αυτό είναι το μόνο που θα πρέπει να συζητάμε. Η στρατηγική της Frontex έχει εξαντλήσει τα όρια της. Δεν είναι πρόβλημα ασφάλειας, δεν είναι μόνο πρόβλημα ανθρωπιστικής βοήθειας. Είναι ένα πρόβλημα συνολικής ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής. Ευθύνη φέρουν όλα τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Αυτό θα πρέπει να συζητάμε τώρα και όχι πώς θα περιορίσουμε τις περικοπές ή τι θα γίνει το ΕΦΣΙ και ορίζον 2020 και ξέρω εγώ η διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη. Αλλά πώς θα διατηρηθούν στο σύνολό τους τα προγράμματα και πώς θα χρησιμοποιήσουμε το περιθώριο που έχουμε φέτος και του χρόνου από τον προπολογισμό ε, και προς τα εκεί θα πρέπει να κινηθούμε και το Κοινοβούλιο και το σύνολο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Έτσι θα δείξουμε την έγκλη, το κύρος μας ε, και ότι μας απασχολεί η συνέχιση της ευρωπαϊκής οικοδόμησης και ολοκλήρωσης ε, που διακυβεύεται όσο ποτέ αυτό τον καιρό αυτές τις μέρες και τις εβδομάδες. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι. Βεβαίως θα δοθεί ευρωπαϊκή απάντηση στη μετανάστευση αλίμονο και θα πρέπει αυτό να βρει και αντανάκλαση στο προπολογισμό του 2016. Δεν ξέρω αν θέλουν το λόγο οι συγητές, ο κύριο Φερνάντε πρώτο ή ο κύριο Δεπρέ, όποιο θέλει, για κάποια σχόλια. Ο κύριος Δεπρέ. Σας ρώτησα αν θέλετε να πάρετε το λόγο για να κλείσετε. Όχι, δεν είναι αναγκαίο. Ωραία, μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι η παρουσίαση από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον ορίζοντα 2020 και τη διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη, το πρόγραμμα COSME και την ε, ε, πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Η Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού θα κάνει αυτή την παρουσίαση και στη συνέχεια καλούνται τα μέλη της Επιτροπής μας να τοποθετηθούν. Και τέλος, δεν ξέρω αν υπάρχουν ειδικέ ερωτήσεις από πλευρά σας. Θα απαντήσει η αρμόδια Γενική Διεύθυνση ε, που είναι αρμόδια για τη διαχείριση των προγραμμάτων αυτών και παρίσταται επίσης. Ο διευθυντή κύριο Πρέζα θα μας κάνει λοιπόν τη παρουσίαση από πλευρά Γενικής διεύθυνση προπολογισμού. Παρακαλώ. Uh, thank Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα σας δώσω μία επισκόπηση της, ε, σχετικά με την πρόοδο στην εφαρμογή των προγραμμάτων που αναφέρετε και θα ήθελα να σας πω ότι οι συνάδελφοι από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση είναι εδώ στη διάθεσή σας για να απαντήσουν σε ενδεχόμενα ερωτήματα που θα έχετε για ζητήματα που θα αναφερθούν στην, ε, στην παρουσίαση. Έχουμε λοιπόν ε, την παρουσίαση με τις διαφάνειες. Είναι πυκνές ε, οι διαφάνειες, θα τις διατρέξω εντάχυν. Και φυσικά είμαι ανοιχτός για περαιτέρω συζητήσεις και ερωτήσεις στη συνέχεια. Ένας κατάλογος επισκόπησης. Δεν ξέρω αν φαίνεται στον πίνακα. Έχετε όμως και την ε, γραπτή το έγγραφο. Τι δείχνει λοιπόν αυτός ο πίνακας για τα τέσσερα προγράμματα για την εφαρμογή του 2014. Πού βρισκόμαστε επίσης το 2015 σε σχέση με το προηγούμενο έτος την ίδια ημερομηνία και στη συνέχεια το ε, επίπεδο των αναλήψεων υποχρεώσεων που έχουν γίνει στον προπολογισμό για το 2016. Έτσι λοιπόν ε, αποκτάτε μια ιδέα για το που βρισκόμαστε. Το βασικό μήνυμα το οποίο προκύπτει από τον πίνακα λοιπόν αυτό είναι ότι, ότι η ταχύτητα εφαρμογή το 2015 επιταχύνθηκε για όλα τα προγράμματα. Και εστιάζομαι ιδιαίτερως ε, στις ε, αναλήψεις υποχρεώσεων σήμερα γενικότερα. Για όλα τα προγράμματα λοιπόν είμαστε πάνω από το επίπεδο της αναλήψη υποχρεώσεων σε σχέση με πριν από ένα έτος, τον Αύγουστο του περσινού έτους. Να τονίσω ότι το 2014, παρά το γεγονό ότι υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις στην έγκριση της ε, νομικής βάσης και αντιμετωπίσαμε δυσκολίες κατά την εκκίνηση, όλα τα προγράμματα σε τελική ανάλυση εφαρμόστηκαν κατά 100%. Η πρόβλεψη τώρα από πλευράς της υπηρεσίας ε, της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής βάσει των προγνωστικών στοιχείων είναι ότι όλα αυτά τα προγράμματα θα έχουν εφαρμοστεί στα τέλη του 2015. Αν περάσουμε λοιπόν τώρα στην επόμενη διαφάνεια τη βλέπουμε. Εδώ σκοπός μας είναι να σας παρουσιάσουμε μεμονωμένα κατά πρόγραμμα τη διαδικασία της εφαρμογής, η οποία μετά την ε, πρόβλεψη στον προϋπολογισμό ζητείται προτάσεις, ε, γίνεται μια επιλογή, ε, μια προχρηματοδότηση και ενδιάμεσες πληρωμές για τον ορίζοντα 20. Έχουμε προτάσεις, μάλλον η έκκληση για υποβολή προτάσεων έχουν, ε, ανέρχονται πλέον στα 16 δισεκατομμύρια. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ποσοστό των χρηματοδότησης στα πλαίσια του ορίζοντα 2020. Η διαδικασία και η εφαρμογή των προγραμμάτων έχει ξεκινήσει. Και αυτό, μάλλον οι, ε, προτάσεις που ζητούνται είναι πολύ πιο πάνω από το επίπεδο των, ε, ε πάνω από την ανάλυση πληρωμών, από τις πιστώσεις. Και τώρα λοιπόν βλέπουμε ότι έχουμε πάνω από 37.000 προτάσεις τις οποίες έχει λάβει η Επιτροπή. Και ε, με 70 δισεκατομμύρια σύμβολοι από τον προπολογισμό. Και το βασικό κριτήριο για την επιλογή των ε, προγραμμάτων των έργων είναι η αριστεία. Έχουμε 4.819 προτάσεις οι οποίες τελικά επιλέχθηκαν. 8,5 δισεκατομμύρια για τον ορίζοντα 2020 έως τώρα λοιπόν. Αυτό σε σχετικούς όρους μας δίνει 13% ποσοστό επιτυχίας των προτάσεων που έχουν επιλεχθεί σε σχέση με αυτές που λάβαμε. Οι υπόλοιπε προτάσεις δε έχουν όλες δημοσιευτεί και όλες ε, οι πιστώσεις θα γίνουν μέχρι το τέλος του 2015. Στον ορίζοντα 2020 έχουμε και ε, χρήματα οικονομικά μέσα, τα οποία τα διαχειρίζεται η ΕΤΕΠ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Αυτό θα επιτρέψει χρηματοδότηση 3,3 δισεκατομμύρια με ευρωπαϊκή συμμετοχή μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και μέσω 2,3 εκατομμυρίων, 2,3 εκατομμυρίων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Και σύμφωνα με τη μελέτη του Ευρωπαϊκού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η εφαρμογή των χρηματοοικονομικών μέσων έρευνας προχωράει πολύ καλά. Και θα υπάρξει μέγιστη απορρόφηση στην ε, περίοδο που καλύπτουν οι αναλήψεις υποχρεώσεων για τα οικονομικά λοιπόν ε, μέσα για τον ορίζοντα 2020 είμαστε σε καλό δρόμο. Να περάσουμε τώρα λίγο γρήγορα στο κόσμο. Ένα πρόγραμμα που αποσκοπεί στις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εδώ έχουμε ε, έλεγχο και χρηματοδότηση. Έχουμε διάφορα επίπεδα χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχά, έχουμε το Enterprise Europe Network, το δίκτυο ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Εδώ έχουμε ε, δύο διαδικασίε πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014. Επιλεφθήκαν 94 όμιλοι που περιλαμβάνουν 559 οργανώσεις και τα 28 κράτη-μέλη καλύπτονται στη... σε ό,τι αφορά τα επιλεγμένα αυτά, στους επιλεγμένους αυτούς ομίλους. Και περίπου 90% του προϋπολογισμού που είχε προβλεφθεί έχει εκχωρηθεί. Τα υπόλοιπα λοιπόν ε, κατά πάσα πιθανότητα θα εκχωρηθούν μέχρι τέλη του έτους. Άρα είμαστε σε καλό ρυθμό. Ένα άλλο στοιχείο του κόσμου είναι το Εράσμου για τους νέους επιχειρηματίες. Ε, είχαμε δύο προσκλήσεις υποβολής προτάσεων το 2014 και το 2015. Στην πρώτη φάση λάβαμε 111 προτάσεις και 15 έργα επιλέχθηκαν. τα στοιχεία για την ε, πρόσκληση υποβολή προτάσεων το 2015 είναι τα εξή. 105 προτάσεις κατατέθηκαν και η αξιολόγηση τώρα βρίσκεται στη φάση της ε, τελικής διαμόρφωσης. Εδώ λοιπόν αναφέρουμε ότι η εφαρμογή ακολουθεί το πρόγραμμα, το χρονοδιάγραμμα. Αντίστοιχα είναι τα πράγματα και για τα χρηματοοικονομικά μέσα, τα οποία περιλαμβάνονται στο κόσμο. Έχουμε το Equity Facility for Growth που δίνει αντεγγύησεις για α, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τη χρηματοδότησή τους και εδώ έχουμε επίσης και την ε, διευκόλυνση για τις εγγύησεις. Στο Equity Facility for Growth πρέπει να γίνει μια μελέτη δεύτερος επιμέλειας από τους διαμεσολαβητές και η επιλογή θα ξεκινήσει στα τέλη του Και τότε θα αναπτύξει τα χειρισμήτα για την, ε, το LGF, το μηχανισμό δανειοδότησης, loan guarantee. Εδώ έχουμε μεγάλη, μεγάλο ενδιαφέρον από τις μικρές ε, επιχειρήσεις και οποιαδήποτε έλλειψη πόρων θα καλυφθεί από το το 2015-2017. Και το συντομότερο δυνατό λοιπόν θα χρησιμοποιηθούν οι πόροι του κόσμου στη συνέχεια. Και εδώ λοιπόν η εφαρμογή ακολουθεί το πρόγραμμα. Περνώντα λοιπόν τώρα στην διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη, Connecting Europe Facility. Εδώ η εφαρμογή και ο τρόπος εφαρμογής μάλλον είναι διαφορετικός. Γιατί το μεγάλο το τμήμα του Connecting Europe Facility περιλαμβάνει ένα πολυετές πρόγραμμα που καλύπτει επταετή περίοδο, την επταετή περίοδο του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Μέσω των πολυετών αυτών προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων, το αντίστοιχο τμήμα του προϋπολογισμού για τα 7 έτη είναι ήδη προκαθορισμένο και ως εκ τούτου σε κάθε ετήσια μερίδα που εγκρίνεται οι πόροι χωρούνται στα επιλεγμένα έργα που έχουν επιλεχθεί μέσα από την πολιετή πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Τα ποσά δε που έχουν ήδη εκχωρηθεί. Ανέρχονται 14,6 δισεκατομμύρια για, την μεταφορά, για τις μεταφορές ε, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών πόρων. Έχουμε περίπου 2 δισεκατομμύρια για την ενέργεια και 320 εκατομμύρια για τον παράγοντα το τμήμα των τηλεπικοινωνιών του Connecting Europe Facility. Να αναφέρω ότι σε κάποια από τα τρία σκέλη αυτά υπάρχουν και ετήσια προγράμματα, ετήσια έργα τα οποία περιλαμβάνονται στην πρόσκληση υποβολή προτάσεων. Αν κοιτάξουμε λοιπόν ε, επιγραμματικά τους τρεις αυτούς ε, κλάδους, ε, Connecting Europe Facility, μεταφορές. Έχουμε τέσσερα πολιετή και τέσσερις μάλλον πολιτικές διαδικασίες και μία ετήσια διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων η επιλογή ολοκληρώθηκε φέτος τον Ιούλιο. Και το αποτέλεσμα λοιπόν είναι το εξή. Έχουμε λάβει 681 προτάσεις ύψους 33, 33 δισεκατομμυρίων. 13 δισεκατομμύρια εκχωρήθηκαν τελικά σε 276 έργα Στις 276 προτάσεις. Στη φάση λοιπόν αυτή υπογράφονται οι μεμονωμένες ε, συμβάσεις με μια προχρηματοδότηση που προβλέπεται από τώρα μέχρι τα τέλη του έτους. Πώς έχει η κατάσταση σε ό,τι αφορά την ενέργεια, το σκέλος της ενέργειας από το Connecting Europe Facility. Έγινε μια πρώτη διαδικασία πρόσκλησης υποβολή προτάσεων το 2014, ετής και άλλες ε, δύο διαδικασίες το 2015. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του 2014, το αποτέλεσμα είναι ότι εκχωρήθηκαν 647 εκατομμύρια σε 34 έργα. Και για τις δύο διαδικασίες του 2015, 150 εκατομμύρια εκχωρήθηκαν σε 20 έργα. Η τρίτη διαδικασία πρόσκληση υποβολών προτάσεων, προκήρυξη, θα εκχωρήσει τον υπόλοιπο προπολογισμό. Τον υπόλοιπο για το 2015. Τέλος. Από πλευρά του Connecting Europe Facility στο σκέλος των τηλεπικοινωνιών. Τρεις προκηρύξεις. 28 εκατομμύρια για έργα τηλεπικοινωνιών το 2014 Οκτώ τέτοιες προκηρύξεις ε, θα γίνουν τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του τρέχοντος έτους, συνολικού ποσού ύψους 46 εκατομμυρίων. Επίσης έχουμε και ένα σκέλος ε, χρηματοοικονομικών μέσων. Εδώ η διαδικασία διαρκεί πιο πολύ από τις επιδοτήσεις Ωστόσο, η συμφωνία ανάθεση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υπεγράφει τι 22 Ιουλίου του 2015 και οι υφιστάμενε ε, διαδικασίες στο Project Bonds Pilot και στο Loan Guarantee έχουν συγχωνευτεί με το νέο μέσο χρέωσης. Τέλος, να δούμε την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Θα σας υπενθυμίσω ότι το 2014 και 2015 στους ε, αντίστοιχους προϋπολογισμούς εκχωρήθηκαν 3,2 δισεκατομμύρια και μάλιστα ε, βαρό για τα δύο έτη αυτά. Ανταποκρινόμενοι φυσικά στα υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων. Και εδώ θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι τουλάχιστον αντίστοιχο ποσό 3,2 δισεκατομμυρίων θα κινητοποιηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Συνολικά δηλαδή φτάνουμε στα 6,4 δισεκατομμύρια σε ό,τι αφορά τις αναλήψεις υποχρεώσεων του 2014 και 2015. Οι αναλήψεις υποχρεώσεων έχουν γίνει με εξαίρεση ενός λειτουργικού προγράμματος το οποίο θα ολοκληρωθεί στην επεξεργασία του το Σεπτέμβριο και εκεί θα γίνει η ανάληψη υποχρεώσεων και μετά την αλλαγή της αρχικής πρότασης σε ό,τι αφορά την προχρηματοδότηση το 30% του πακέτου, του φακέλου θα χορηγηθεί υπό μορφή προχρηματοδότηση το 2015. Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή, επιτόπια εφαρμογή, ήταν αρκετά αργή η εκκίνηση το 2014, αλλά τώρα βλέπουμε ότι επιταχύνει το πρόγραμμα. Οι δικαιούχοι του προγράμματος αναμένεται ότι θα φτάσουν τους 900.000 το 2016 και τα επόμενα δύο έτη θα προσθεθεί ένα εκατομμύριο επιπλέον σε ό,τι αφορά τους δικαιούχους του προγράμματος. Ως εκ του η εφαρμογή θα διαμοιραστεί μεταξύ του 2015, του τρέχοντος έτου, έτους, μέχρι και το 2018. Δεν θα υπάρχει λοιπόν ασυνέχεια μετά το 2015, δεν θα υπάρξει διακοπή της εφαρμογής. Ένα τελευταίο σημείο για την πρωτοβουλία απασχόληση των νέων από πλευρά των πληρωμών τώρα. Ένα τρίτο περίπου των συνολικών ποσών που περιλαμβάνονται στις αναλήψεις υποχρεώσεων θα δοθεί το 2015, άλλο ένα τρίτο το 2016 και το υπόλοιπο μετά το 2016. Και για να σας προλάβω στην ενδεχόμενη ερώτηση που θα έχετε, τι θα γίνει μετά το 2015 με την πρωτοβουλία απασχόλησης των νέων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τις πρώτες ε, αξιολογήσεις τις οποίες ε, αναμένουμε στα τέλη του έτους και στα πλαίσια της ενδιάμεσης αναθεώρησης του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου θα αξιολογηθεί κατά πόσο η παράταση της πρωτοβουλίας ε, αυτής ε, είναι επιθυμητή βάσει των, απο... επιτευγμάτων, των αποτελεσμάτων. Θα σταματήσω κάπου εδώ. Το βασικό μήνυμα είναι ότι συνολικά και στα τέσσερα προγράμματα η εφαρμογή πηγαίνει καλά. Και ακολουθεί το χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρέζα. Δεν ξέρω αν έχετε ερωτήσεις, παρατηρήσεις. Συνάδελφοι, κύριος Φερνάντες, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την παρουσίαση. Ευχαριστώ πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκτέλεση. Μπορείτε να τα πείτε αυτά και στο Συμβούλιο παρακαλώ πολύ, γιατί αν δεν έχει την ίδια πληροφόρηση και το Συμβούλιο, ε, θα συνεχίσει τις περικοπές. Εάν λάβει αυτή την πληροφόρηση μπορεί να το χωνέψει και να σταματήσει τις περικοπές. Γιατί ένα από τα κριτήρια που επικαλείται το Συμβούλιο είναι η απορροφητικότητα και η εκτέλεση. Μπορείτε παρακαλώ το συντομότερο να τα διαβιβάσετε αυτά στο Συμβούλιο για να καταλάβει τι γίνεται για να αναθεωρήσει τη θέση του, διότι η τελική ε, ψηφοφορία θα γίνει βάσει της ανάλυσης ε, του Κορεπέρ, αύριο δηλαδή. Θα ήθελα λοιπόν να πω απλώς ότι σε ό,τι αφορά την εκτέλεση ε, του ορίζοντα 2020, του κόσμε, ε, Τη ευκόλυσης συνδέοντα στην Ευρώπη, όλα αυτά τα προγράμματα δείχνουν και μάλιστα με τρόπο επαρκή ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε δίκιο στη θέση που έλαβε. ζήτησε οπωσδήποτε ενίσχυση και διατήρηση όλων αυτών των πιστώσεων, διότι η εκτέλεσή τους ε, ανταποκρίνεται απολύτως όχι απλώς ε, στις προσδοκίες και στις φιλοδοξίες, αλλά και στους ίδιους τους στόχους, ε, μάλιστα 100%. Οπότε δεν καταλαβαίνουμε γιατί εξακολουθεί το Συμβούλιο να εμένει στις περικοπές αυτών ακριβώς των κονδυλίων που είναι εκείνα που απορροφούν το περισσότερο. Δεν ξέρω, μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ε, απαντήσει σε αυτό ή να μας δώσει επιχειρήματα για να μας βοηθήσουν να πείσουμε εμεί στο Συμβούλιο για το πόσο μεγάλη σημασία έχουν αυτά τα προγράμματα. Αν κατάλαβα καλά, ε, υπάρχουν ορισμένες επιστώσεις του κόσμου που δεν έφτασαν, χρειάστηκαν για τα χρηματοδοτικά μέσα επιπλέον ε, κονδύλια. Και αφού είναι σημαντικό λοιπόν αυτό το πρόγραμμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν θα πρέπει να αυξηθεί η πρικοδότησή του. Και σε ό,τι αφορά την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, κοιτάξτε πώς είναι οι άνεργοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν μειωθεί οι θέσεις εργασίας. Για μένα είναι προφανές και αυτονόητο ότι πρέπει να διατηρηθεί αυτή η πρωτοβουλία. Για ποιο λόγο καθυστέρησε η εφαρμογή και η εκτέλεσή της στα κράτη-μέλη. Υπάρχουν κράτη όπου παρατηρείται τεράστια καθυστέρηση και κατάφορη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2016 θα ζητήσει να δοθεί απαραίτητη άδεια για να συνεχιστεί η πρωτοβουλία. Θέλω να μάθω όμως και τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για ποιο λόγο καθυστέρησε η υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων στα κράτη-μέλη. Για να έχουμε και εμείς επιχειρήματα, για να επιμείνουμε και να πιέσουμε το Συμβούλιο για τη σημασία ακριβώς αυτής της πρωτοβουλίας. Γιατί ξέρετε ότι η απασχόληση των νέων είναι για μας προτεραιότητα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φερνάντες. Η κυρία Γκουαρια Σάμπαλ που είναι η συγκήτρια του προπολογισμού για το 2015. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Το πρώτο που πρέπει να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να διαβιβάσει τα στοιχεία αυτά στο Συμβόλιο. Έχει απολύτω δίκιο ο κύριο Φερνάντε. Στη δική μα Επιτροπή, όποτε λέμε ότι δεν φτάνουν τα λεφτά, ότι τα προγράμματα υποχρηματοδοτούνται, πάντα μας απαντούν ότι οι περικοπές που κάνει το Συμβούλιο είναι γιατί δεν απορροφούνται τα κονδύλια, γιατί τα λεφτά περισσεύουν και τα λοιπά και δεν τα κάνουμε τίποτα. Είναι πολύ εύγλωτα τα στοιχεία, έχει πολλά έργα η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι και χρήσιμα και υλοποιούνται και απορροφούνται. Όταν εμείς από τη δική μας Επιτροπή ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έρθει να μας παρουσιάσει την εκτέλεση αυτών των προγραμμάτων, ε, το κάναμε και εν ώψη της προετοιμασίας του προϋπολογισμού του 2016. Γιατί δεν θα ήταν λογικό αν δούμε ότι δεν είναι καλή εκτέλεση των προγραμμάτων ή καθυστερούν, δεν έχει νόημα λέγω να ζητάμε περισσότερα λεφτά με όλες αυτές τις προτεραιότητες που έχουμε και τις κατεπίγουσες ανάγκες ε, που πρέπει να καλύψουμε. Είναι γεγονός όμως ότι τα στοιχεία που μας δίνονται και τα αριθμητικά, τα περισσότερα, ε, είναι σε καλό δρόμο, έχουν αποκτήσει τώρα μία ε, πορεία στις δικές μας τροπολογίες μπορεί να χρειαστεί να ζητήσουμε περισσότερα χρήματα για τον ορίζοντα 2020 και το ΣΕΦ, γιατί έπεσαν θύματα στο βωμό του ΕΦΣΙ, του Ταμείου Στρατηγικών Επενθύσεων. Έχω λοιπόν δύο ερωτήσεις. Για τον κόσμο πρώτα. Έχετε ένα πίνακα εδώ που λέτε για το μηχανισμό εγκυοδότησης των δανείων. Λέτε ότι υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση από ότι ε, προσφορά. Προς το παρόν καλύπτεται αυτό από το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, ε, αλλά ε, δεν έχω καταλάβει τι γίνεται ακριβώς με τα αριθμητικά στοιχεία. Και σε ό,τι αφορά την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, καθυστέρησε πολύ να κινήσει. Τα κράτη υπέβαλαν τα επιχειρησιακά του σχέδια αργά. Τα αριθμητικά στοιχεία δεν είναι καλά, παρατηρούνται καθυστερήσεις και είναι επίγον. Από το 2013 μας αποσχολεί αυτή η πρωτοβουλία που αποφασίστηκε και μέχρι το 2016 δεν θα έχει εφαρμοστεί καλά. Ε, ε, αυτή είναι μία ερώτηση. Και η δεύτερη, και αν έχετε στοιχεία να μου τα δώσετε από την Κομισιόν, γιατί φτάσανε στα αυτιά μου σχόλια που λένε ότι εκεί που έχει αρχίσει η ε, εφαρμογή της πρωτοβουλίας δεν έχει δώσει τα απαραίτητα και τα επιθυμητά αποτελέσματα. Δηλαδή δεν μπαίνουν οι νέοι στην αγορά εργασίας, κάνουν ασκήσεις, στάζ, πρακτικές κτλ. Αλλά αυτό στρεβλώνει ε, την εργασία, δεν δημιουργεί θέσεις εργασίας, απλώς ε, δημιουργεί επισφαλής και κακής ποιότητας θέσεις εργασίας και με κακές αμοιβέ για μικρό χρονικό διάστημα. Το σκέφτεστε αυτό, σας έχει απασχολήσει και πώς μπορεί να λυθεί. Πώς μπορεί να βελτιωθεί και κυρίως τι θα γίνει στο μέλλον. Διότι το 14 και το 15 ε, είχαμε κάποια χρήματα, για το 16 δεν υπάρχουν ε, δεσμεύσεις, ε, δηλαδή κονδύλια ανάληψη υποχρεώσεων και για το 17 βλέπουμε. Και μετά θα μας μένουν τρία χρόνια μέχρι το 2020 και η ανεργία των νέων θα έχει ξεφτήσει στο 50%. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν θέλει κανείς άλλο το λόγο. Αν όχι, τώρα θα δώσω το λόγο πάλι στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στους άλλους συναδέλφους για τα προγράμματα COSME και για την απασχόληση των νέων για να απαντήσουν στις ειδικότερε ερωτήσεις των βουλευτών. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα απαντήσω στη γενική ερώτηση του κυρίου Φερνάντες και της κυρίας Γκαρδιαθάβαλ. για αυτά τα, αν θα δώσουμε αυτά νούμερα για την υλοποίηση στο Συμβούλιο. Ξέρετε, η απάντηση μου είναι εξή. Η Επιτροπή κάθε εβδομάδα στέλνει τους αριθμούς ε, για την υλοποίηση σε αναλήψη υποχρεώσεων ε, και πληρωμές και στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Το Συμβούλιο αιτιολόγησε τις ε, περικοπές ε, λέγοντας ότι είδε την εφαρμογή, αυτό είναι το επιχείρημα τους, είδε το βαθμό εφαρμογής τον Ιούνιο και μετά βάσει αυτού υποθέτω ποια θα είναι η κατάσταση το 2015, τι θα παραμείνει και κάνουμε τις αναλόγες περίκοπες. Φυσικά τον Ιούνιο δεν έχει ακόμα εκτελεστεί όλος ο προπολογισμό. Διότι ξέρετε υπάρχει μια διαδοχή, μια λιλουχία πραγμάτων, ε, προκηρύξεις, επιλογή, ε, επεξεργασία των στοιχείων, ε, σύναψη της σύμβασης πριν εκταμιευθούν τα χρήματα. Ουσιαστικά τα νούμερα τώρα, το, στα τέλη Αυγούστου, αντιστρέφουν, δίνουν άλλη εικόνα για την κατάσταση εφαρμογής πολλών από αυτά τα κονδύλια. Οπότε η λογική που χρησιμοποιήθηκε για τις περικοπές λογικά του Συμβουλίου θα έπρεπε να αντιστραφεί. Ε, αλλιώς εντάξει, αυτό δεν θα γίνει έτσι αυτόματα. Αν μου επιτρέπετε να δώσω το λόγο στην κυρία Σούκοβα που κάθεται δίπλα μου για την πρωτοβουλία απασχόληση των νέων και στην κυρία Νέμεν για το κόσμο. και την κυρία Ρέτε. συγγνώμη. Λοιπόν, έχετε το λόγο για συγκεκριμένες ερωτήσεις για τις καθυστερήσεις, τα αποτελέσματα, για τους τύπους ε, θέσεων εργασία που δημιουργήθηκαν, για την κατάσταση επιμέρους κράτη-μέλη, ερωτήσεις που έγιναν από τα μέλη μας. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ γιατί είναι σημαντικό και για την Κομισιόν να φροντίσει να υλοποιεί ποιοτικά έργα που υποστηρίζουν πραγματικά την απασχόληση των νέων στο μέλλον. Μπορώ να αιτιολογήσω την έλλειψη καλών πληροφοριών, αξιόπιστων πληροφοριών ε, και τυχόν αποτελεσμάτων σε ορισμένα κράτη-μέλη που ε, έκαναν το πρόγραμμα αυτό της απασχόλησης των νέων ε, τόσο περίπλοκο που χρειάστηκε χρόνος για να υιοθετηθεί και για να αξιοποιηθούν τα χρήματα που υπήρχαν διαθέσιμα βάσει του κονδυλίου και να δοθούν αυτά τα χρήματα στις περιφέρειες. Η υιοθέτηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων συνέχισε το 2015 και συνεχίζει απαωμένη ένα με στοιχείο ε, για την απασχόληση των νέων που δεν έχει ακόμα υιοθετηθεί αλλά πιστεύουμε ότι μεσα στα τέλη του Σεπτεμβρίου και τα 34 επιχειρησιακά προγράμματα θα έχουν υλοποιηθεί, θα έχουν υιοθετηθεί. Η υιοθέτηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων δεν είναι παρά η αρχή της υλοποίησης, ε, της πραγματοποίησης των δαπανών. Τα κριτήρια επιλογής που έχουν συμφωνηθεί με τις Επιτροπές Παρακολούθησης δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί σε πολλά κράτη-μέλη. Οι μεγαλύτεροι δικαιού, δικαιούχοι δυστυχώς είναι αυτά τα κράτη-μέλη. Σε ορισμένε περιπτώσει έχουμε αυτή τη στιγμή οργανώσει συναντήσει τον Σεπτέμβριο για να οριστικοποιηθεί η διαδικασία ο καθορισμού των κριτηρίων και για να διασφαλίσουμε την επιτάχυνση τη υλοποίηση των προγραμμάτων. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο απαραίτητο για την υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της δυνατότητας των δημόσιων υπηρεσιών και των ενδιάμεσων οργάνων που συμμετέχουν στην όλη διαδικασία να έρθουν σε επαφή με ε, ανθρώπους ανέργους ε, και που δεν απασχολούνται και που δεν σπουδάζουν ε, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα μέσα αυτά λειτουργούν σωστά και επιλέγουν σωστά αντιμετωπίζετε τις ανάγκες των νέων. Ακόμα δεν έχουμε ορίσει τις αρχές για τα επιχειρησιακά προγράμματα που αποτελεί προϋπόθεση για τα κράτη-μέλη ώστε να στείλουν αιτήσει πληρωμών στην Κομισιόν σε σχέση με την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Δυστυχώς, στα κράτη-μέλη παρατηρήθηκαν πολλές καθυστερήσεις όσον αφορά την υλοποίηση των προγραμμάτων, τεχνικές και διοικητικές. Μέσω των συναντήσεων ε, της επιτροπής, των Επιτροπών Παρακολούθησης που συμμετέχουν ε, ε, συναδέλφοι από την Επιτροπή, πιστεύουμε ότι ακολουθούμε αυτή τη στιγμή το χρονοδιάγραμμα και ελπίζουμε σε μια καλύτερη εκτίμηση των αποτελεσμάτων προς τα τέλη του έτους. Φυσικά αναζητούμε ποιοτικά μέτρα και μεταρρυθμίσεις και θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο η δαπάρη των 6,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων στην Ευρώπη. Τα επιχειρησιακά προγράμματα που υιοθετήθηκαν μέχρι στιγμής, τα περισσότερα δηλαδή, δείχνουν ότι τα κράτη-μέλη, τα οποία δεν είναι επιλέξιμα για την πρωτοβουλία απασχόληση των νέων, έχουν ήδη προγραμματίσει δράση και μέτρα για να αντιμετωπίσουν την ανεργία των νέων. Το συνολικό κονδύλιο αυτή τη στιγμή είναι 12,7 δις ευρώ αντί για 6,4 για μέτρα που παρέχουν πρόσβαση σε νέους ανέργους ε, και σε νέες δυνατότητες. Μιλάμε λοιπόν για υψηλότερο νούμερο. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η πρόβλεψη στο, η διάταξη στο άρθρο 14 του κανονισμού του πολιτούς ε, το πλαισίου, δημοσιονομικού πλαισίου λέει ότι του χρόνου ο προπολογισμό θα δώσει προτεραιότητα σε δράσεις απασχόλησης των νέων και ελπίζουμε ότι θα συνεχιστούν οι δεσμεύσει του προηγούμενου κοινοβουλίου για να συνεχιστεί η προσπάθεια σε αυτόν τον τομέα με περαιτέρω χρηματοδότηση, τη συνολική χρηματοδότηση για την αρρωγή προς ε, ενίσχυση των ε, άνω των 5 εκατομμυρίων νέων ενέργων στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα για συγκεκριμένες απαντήσεις για το κόσμο, η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξη ο, αναπληρωτή αναπληρωτής τμήματάρχης Νάιμαν. Yes, thank you very much. Συγγνώμη, ή. Ε, όντως, ε, ε, τα δύο αυτά προγράμματα είχαν τεράστια ζήτηση το κόσμο και η εγγύηση για τη δανειοδότηση και φυσικά υπερεύησαν τα ποσά που είχαμε στη διάθεσή μας. Όπως είπε και ο κύριος Πρέσα προς το παρόν, χρησιμοποιούμε τη χρηματοδότηση από το Αμείο Στρατηγικών Επενδύσεων για εμπροστοβαρή καταβολή μέχρι τα τέλη του 2017 για να καλύψουμε τη ζήτηση που μας κατακλίζει. Μετά το 2017 θα έχουμε πρόβλημα, το 2018 όπου δεν θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα της εμπροστοβαρούς καταβολής. Και βεβαίως έχουμε συζητήσει αυτά τα θέματα σε πολύ στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων που λέει ότι για το 2018 θα χρειαστούμε 100 εκατομμύρια και στη συνέχεια 200 ε, ετησίως για το 2019 και το 2020. 200 εκατομμύρια επιπλέον. Αυτά θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας ε, κατά την αναθεώρηση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Um, Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Δεν ξέρω, θέλει κανείς να απαντήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Πρέστα, τα έχετε να προσθέσετε. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να δώσω το λόγο σε μια συνάδελφο για να προσθέσει για το κόσμο, την κυρία Ρούτα. Ευχαριστώ πολύ. Μάι Ρούτα, από τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας. Ο κύριος Φερνάντες και ε, Κάποιος άλλος συνάδελφος, η κυρία Καρδιασάβρου, ρώτησε τι γίνεται με την ε, απορρόφηση ε, για την ε, απασχόληση των νέων. Για τον ορίζοντα 2020 και στο πρόγραμμα πλαίσιο παριθμών 7 το προηγούμενο είχαν 100% απορρόφηση κάθε χρόνο, χρόνο με το χρόνο. Δεν υπάρχει λόγος να αμφισβητήσουμε αυτό το γεγονός και φέτος θα συμβεί και στην ανάληψη υποχρέωσεων και στις πιστώσεις πληρωμών αρκεί το Συμβούλιο να δει τα στοιχεία. Αν έχει τα στοιχεία του Ιουνίου, είναι πολύ νωρί. Τέλη του έτου πρέπει να κοιτάζει τα στοιχεία το Συμβόλιο. Το δεύτερο που ρώτησε ο κύριο Φερνάντε είχε να κάνει με του λόγου για του οποίου χρειάζεται αυτό ο προπολογισμό. Θέλω να θέσω υπόψη σα ε, μια πολύ σημαντική τάση που παρατηρούμε αυτό τον καιρό. Σε σύγκριση με το προηγούμενο πρόγραμμα, ε, το πρόγραμμα πλαίσιο το 7ο, ε, για την καινοτομία και την έρευνα σήμερα ε, είναι ε, πολύ υψηλότερη η ζήτηση. Και ακόμα και τα εξαιρετικά προγράμματα δεν μπορούμε να τα χρηματοδοτούμε. Αυτά που βαθμολογούνται ως εξαιρετικά στο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα. Και μόλις 20% ε, καλύψαμε και αυτό έχει γίνει στο μεταξύ 13% και σε ορισμένα διαγωνισμούς που έχουν να κάνει με έρευνα για την υγεία είναι στο 4%. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πάρα πολύ καλά προγράμματα που βαθμολογούνται και αξιολογούνται ως εξαιρετικά και δεν μπορούν να βρουν χρηματοδότηση. Και εδώ μιλάμε για την καινοτομία, η Ευρώπη χρειάζεται οπωσδήποτε. Γι' αυτό θα πρέπει να πιέσουμε για μεγαλύτερη χρηματοδότηση και υψηλότερη ακριβώς αυτούς τους τομείς έρευνας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ζητάει κανείς άλλος ε, το λόγο από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν όχι, θεωρούμε λοιπόν ότι ολοκληρώνεται η συζήτηση για το θέμα αυτό στη σημερινή συζήτηση. Να περάσουμε στο επόμενο σημείο. Ψηφοφορία για την έκθεση του κ. Ντεπρέ και την κατάσταση στην περιοχή της Μεσογείου και την ανάγκη για μια ολιστική προεξέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη μετανάστευση. So we, we start now the, the voting procedure. Να ξεκινήσουμε λοιπόν τις ψηφοφορίες. Ε, στην παραγράφο 1. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παραγράφος 1. Πρωτοπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 1. Ε, τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παραγράφος 2. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 2α. Τροπολογία 7. Υπέρ. Παράγραφος 2. Τροπολογία. Όλες οι τροπολογίες, οι 6, 5 και 4, καταπίπτουν μια και εγκρίθηκε ο συμβιβασμό. Η τροπολογία 7 λοιπόν, υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Παράγραφο 3, συμβιβαστική 2, υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Παράγραφος 4 ή 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 4α, τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παραγραφός 5. Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παραγραφός 5. Τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Παράγραφος 5. Τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Παράγραφος 6. Τροπολογία 16. Υπέρ. Κατά να ελέγξουμε παρακαλώ μέσω της ηλεκτρονικής οδού για την παράγραφο 6, τροπολογία 16, έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Ναι, ψήφισατε όλοι. Ψήφισατε παρακαλώ όλοι. So Yes. The, okay, the, the vote is... Πέρας της So it is rejected. Απορρίπτεται. Όχι απορρίπτεται. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας είναι ξεκάθαρο. Απορρίπτεται. Παράγραφος 7, τροπολογία 17, υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε και πάλι ηλεκτρονικά, παρακαλώ. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Πέρας. Η τροπολογία εγκρίνεται. Παράγραφος 7, τροπολογία 18. Υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά ας το ελέγξουμε παρακαλώ. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Και η τροπολογία απορρίπτεται. Παράγραφο 7. Τροπολογία 19 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 7α. Τροπολογία 20 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 7β 21 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 8α 22 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 9. Τροπολογία 23 υπέρ Κατά. Νομίζω... Α, αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Ας το ελέγξουμε, ας το ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Έναρξη ψηφοφορία. Την 23. Τροπολογία 23. Πέρασε. Απορρίπτεται η παράγραφος 10, 24 τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 10, 25. Καταπίπτει γιατί εγκρίθηκε 24. Η παράγραφος 11, τροπολογία 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα η ψηφοφορία επί του κειμένου όπως τροποποιήθηκε. Με ονομαστική κλίση παρακαλώ. Έναρξη ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 23 ψήφοι υπέρ, 4 κατά, 3 αποχές. Για το επόμενο σημείο στην ημερήσια διατάξη δεν υπάρχουν αιτήσει μεταφορά ούτε από την κυρία Ρελιζαμπάλ, ούτε από την κυρία Χόλμαερ.